Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα ακούσουμε τις επεξηγήσεις ψήφου και γι' αυτό σας ζητώ παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα. Θα ξεκινήσουμε με την έκθεση Κουν. Δέκα φορές χτύπησα και ούτε αυτό αρκεί από ό,τι φαίνεται, γι' αυτό παρακαλώ συνάδελφοι να βγείτε και να κάνετε λίγη ησυχία. Θα ζητήσω το λόγο από τον κύριο Καπούτο να μας δώσει την επεξήγησή του για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο κύριε Καπούτο. Ο κύριος το επαναλαμβάνω, έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε.